δηλώνει ότι αυτές οι δύο έδρες είναι κενές από τις 25 Φεβρουαρίου ε, ενεστώτος έτους. Και τελευταία ανακοίνωση, η υπογραφή των νομικών πράξεων ε, γίνεται, λαμβάνει χώρο μέσα της κανονικής, της συνηθισμένης διαδικασίας. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου και τη Δευτέρα και εγώ θα υπογράψουμε τέσσερις πράξεις δυνάμει το άρθρο 74 ε, το εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σημειώνω ότι θα δημοσιευτούν οι πράξεις στα πρακτικά της ε, τριχούσης συνόδου. Θα δημοσιευθούν στα πρακτικά. Νομοθετικές πράξεις θα δημοσιευθούν αυτές στα πρακτικά. Και πάμε στον καθορισμό του προγράμματος αυτής της εβδομάδας, της συνόδου μας αυτής.